αιτίας. Ίσως να κράτησε πολύ καιρό όμω αυτό. Διαπιστώνω όμω ότι κάποια από τα επιτέματα από το 2016 και μετά σε επίπεδο δημοκρατία επαναχωρούν. Είναι προ συμφέρον όλων οι καλή σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και το καθένα από τα κράτη-μέλη μα. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να επαγρυπνεί ε, και να είναι ενημερωμένη όταν καταδικάζει ανθρώπινα δικαιώματα και παραβίαση του κράτου δικαίου. Αλλά ο διάλογο πρέπει να παραμένει ανοιχτό υπηκοδομητικό σταθερός με αυτήν τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά. Επίσης χρειάζεται στενός διάλογος, ευθυγράμμιση στην εξωτερική πολιτική, πολιτική άμυνας, πολιτική ασφάλειας, επικεντρωνόμενη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ζητήματα στρατιωτικής και στρατηγικής σημασίας. Είναι και η Τουρκία ένα πολύ ε, σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ, ε, της στρατιωτικής αυτής συμμαχίας. Τέλος, ενώ η Τουρκία ε, είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας εμπορικά, με τη Γερμανία στην πρώτη γραμμή, η Τελωνιακή Ένωση εξακολουθεί ε, να μένει στα ίδια. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει η προπαρασκευή για την ε, αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης και στο μέτρο του δυνατού να έχουμε όσο γίνεται πιο σύντομα την επόμενη εντολή. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο ε, ε, Ο κ. Χριστοφόρου θέλει να θέσει ένα ερώτημα όμω. Παρακαλώ, κ. Χριστοφόρου, κίτρινη κάρτα. Στην να αναφέρεται πολλέ φορέ ότι η Τουρκία είναι ένα εταίρο. Ήθελα πραγματικά να μα εξηγήσετε εμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώ εννοούμε και πώ αισθανόμαστε του εταίρου. Εταίροι όπω την Τουρκία που είναι ο πλέον αναξιόπιστο, ο πλέον προκλητικό εταίρο ο οποίο επιτίθεται σε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να ξέρω αν η Τουρκία επι... επιτιθέτων στη Ρουμανία κατά τον ίδιο τρόπο που επιτίθεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αυτή θα ήταν η αντίδρασή σα. Εάν στη Ρουμανία η Τουρκία δεν αναγνώριζε την χώρα ω χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ω μια ανεξάρτητη χώρα όπω δεν αναγνωρίζει την Κύπρο, θα θεωρούσατε την Τουρκία αναξιόπιστον εταίρων που οφείλουμε να συνεχίσουμε να την αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο χωρί να λαμβάνουμε μέτρα και κυρώσει. Okay. Ε, αγαπητέ συνάδελφε, εγώ την Τουρκία δεν τη βλέπω με τα ρουμανικά μάτια. Εδώ είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξετάζω το ρόλο της Τουρκίας από ευρωπαϊκής προοπτικής. Δεν έχει σημασία τι λέτε εσείς ή τι λέω εγώ ή πώς το βλέπω εγώ προσωπικά. Η Τουρκία είναι εκεί, γεωγραφικά είναι εκεί, πολιτικά είναι εκεί, στρατιωτικά είναι εκεί και η Ευρώπη είναι καλό να έχει μια πιο ισχυρή και πιο αποφορτισματική ε, σχέση με την ε, Τουρκία. Είναι πιο ισχυρή έτσι και είναι πιο αδύναμη και κινδυνεύει περισσότερο αν κόψουμε κάθε σχέση με την ε, Τουρκία. Όπως κάνει το ε, ΕΛΚ για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει για την πολιτική του ατζέντα. Δεν συμφωνώ λοιπόν μαζί σας. Ο κύριος Μπέλντερ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούστε, γνωρίζω ότι η έκθεση αυτή έχει κολλήσει σε κάποιο γραφείο ε, από αυτά τα γραφεία που έχουν μεγάλη επιρροή και που χρηματοδοτώνται ε, με μεγάλους προπολογισμούς. 120.000 εργαζόμενοι εκεί εργάζονται. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν κύριε Επίτροπε. Ε, κοιτάξτε την έκθεση του κυρίου Σίβιτς ε, τη μελέτη για τον Ερντογάν. Διαβάστε τα αυτά. Πραγματικά πρέπει να τα διαβάσετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξτάσουν πολύ προσεκτικά το ζήτημα αυτό. Θα έχουμε μια νέα έκθεση από την Κομισιόν σύντομα, διότι είναι πολλές οι παράνομες δραστηριότητε των ε, ε, οξυματούχων του DNET ε, κατασκοπία είναι και μια προσπάθεια καταπολέμησης ε, του αντισημιτισμού ε, υπάρχει το θέμα των μειονοτήτων μιλάμε για την προστασία ηγετών που είναι όμως αντισημίτες ε, χάσαμε λοιπόν μια ευκαιρία να μιλήσουμε καθαρά για το θέμα αυτό και να μην δεχτούμε αυτήν την τροπολογία η Μαριέτε έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ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 Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ετήσια συζήτηση για την πρόοδο της Τουρκίας προς την κατεύθυνση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλο και πιο δύσκολη και πιο επώδυνη. Τώρα έχουμε την έκθεση πρόοδου. Τα τελευταία χρόνια ή τον τελευταίο χρόνο συνέβησαν πάρα πολλά και νομίζω, εντάξει, σωστό ήταν το να διωχθούν ε, οι υπέτοι ε, για το, την απόπειρα πραξικοπήματος, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει και υπεραντίδρυση. Γιατί καταλήξαμε στο να απολύονται εκατοντάδες άνθρωποι, να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα κατά τι τρομοκρατίε, να περιορίζεται η ελευθερία τύπου, ε, κατηγορίες έναντι ε, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως το Σμαν Καβαλά. Σε γενικές γραμμές, οι βασικές αρχές ε, κινδυνεύουν. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η διάκριση των εξουσιών, το κράτος δικαίου, όλα αυτά κινδυνεύουν και αυτά επηρεάζουν την αντιπολίτευση τη γυναίκα σε τους ΛΟΑΔ, ε, τις θρησκευτικέ ενότητες, ε, τους αμύντορες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και πολλούς άλλους και πολλές άλλες μειονότητες. Σχεδόν όλοι στην Τουρκία, είτε ανοιχτά είτε σιωπηρά στην καρδιά τους, γνωρίζουν πολύ καλά τι διαδραματίζεται και φοβούνται το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον φόβος για το τι μπορεί να πάει στραβά. Αυτός ο φόβος έχει παραλύσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μήπως ε, επειδή μας ενδιαφέρει να έχουμε κάπου να πηγαίνουν οι πρόσφυγες ε, αυτό τελικά επισκιάζει τα πάντα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι διακυβεύεται η αξιοπιστία μας και επιμένω τα λόγια μας και οι αρχές μας να έχουν νόημα. Όπως έχουμε προειδοποιήσει και κατά το παρελθόν με την έγκριση του πακέτου συνταγματικών μεταρρυθμίσεων τώρα πλέον έχει εγκατασταθεί ένα προεδρικό σύστημα χωρίς πολλούς ελέγχους και αυτό όχι με αυτά που λέμε εμείς αλλά με όσα λέει η Επιτροπή της Βενετίας. Ε, να συνεχίσουμε ίσως ε, τη σχέση θέσεις μας στο εμπόριο ή ε, για τους πρόσφυγες, αλλά να δουλεύουμε πάντα με την Τουρκία επί τη βάση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επόμενος ομιλητής, Βαλέρο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς έχει συμβεί η εισβολή στο Αφρίμ. Πήγαμε επιτόπου στο Διαμπακύρ και εκεί ε, διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ε, η κοινωνία των πολιτών, υπάρχει ένα δίκτυο ε, το οποίο όμως υποφέρει πάρα πολύ. Και βλέπουμε ότι παραβιάζονται κυρίως ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, συγκεκριμένα κατά την εισβολή στο Αφρίμ. Ε, δεν μπορεί κανείς να πει οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Είναι πολύ δύσκολο να συνεχιστούν βέβαια οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Από την άλλη δεν πρέπει να κλείσουμε τελείως την πόρτα. ομάδες ε, Συρίων και άλλοι ε, τρομοκράτες ε, στη Βόρεια Συρία αυτοί δυστυχώς στηρίζονται πολλές φορές όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι ομάδες των Κούρδων δεν πρέπει να απειλούνται. Είναι εκείνοι οι οποίοι ε, αντιμετωπίζουν το Ισλαμικό κράτος. Η Τουρκία βέβαια θα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Όλα αυτά είναι κατοχυρωμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο κάπως έχουμε κουραστεί να παρακολουθούμε όλες αυτές τις ε, εξελίξεις. Ε, βλέπουμε ότι η απόπειρα πραξικοπήματος ήταν κάτι το οποίο σαφώς και καταδικάζουμε. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ε, συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, οι δημοκρατικές μειονότητες αντιμετωπίζονται εχθρικά. Δεν θέλουμε να παγωθούν οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν κ. Χατζηγεωργιού. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Χάν, κυρία Πύρη, αγαπητοί συνάδελφοι. Ίσως αυτή είναι η τελευταία ουσιαστική μου παρέμβαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενός πολύ φιλόδοξου πειράματος που ανέλαβε ποτέ η ανθρωπότητα. Μιλώντας όμως για την Τουρκία, οφείλω να σας πω και δεν αναφέρεται αυτό μόνο στην Τουρκία, μας λείπει η αλληλεγγύη, αγαπητοί συνάδελφοι, μεταξύ των κρατών μελών και συνακόλουθα δυστυχώς κάποτε και μεταξύ των λαών. Δεν αποτελεί η Κύπρος, προέρχομαι από την Κύπρο και οφείλω να σας πω δύο κουβέντες, δεν αποτελεί η Κύπρος σε αυτή τη συζήτηση κατεχόμενη χώρα. Δεν αποτελεί αναγκαίο βάθος της συζήτησης που ε, λαμβάνει η χώρα σήμερα εδώ. Υπάρχει μια ασάφεια, για να πω το ελάχιστο, στη στάση που έχουμε απέναντι στην Τουρκία και ως κράτη-μέλη αλλά και ως ε, ευρωβουλευτές δεν ξέρουμε τι να πούμε στην τουρκία αλλά την ίδια ώρα η τουρκία ξέρει πολύ καλά τι λέει σε εμά. την ίδια ώρα το ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα ζήτησε τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την χώρα αυτή αλλά την ίδια στιγμή ζητά αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης. είναι σαν να παίρνεις από κάποιον το ψωμί αλλά του δίνεις το φούρνο και το σιτάρι. θεωρώ ότι αυτή είναι μια λανθασμένη προσέγγιση. πρέπει να είμαστε τίμιοι απέναντι στην τουρκία και να ξέρει ακριβώ τι είναι αυτό που ζητούμε από αυτή. Ο κύριο Τσαβούσογλου πρόσφατα, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι αξιωματούχοι, δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, αναφέρονται συχνά πυκνά στην φράση Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε λύση στην Κύπρο. Αυτό εμπεριέχει την βέβαιη τοποθέτηση ότι αναζητούν λύση δύο κρατών. Δεν μπορεί να υπάρξει Κύπριος που θα σηκώσει το στυλό για να υπογράψει λύση δύο κρατών γι' αυτό και το μήνυμα μου και προς τούρκους αξιωματούχους αλλά και ως προς οποιονδήποτε κύπριο είναι ότι πρέπει να ανασχεθεί αμέσως η οποιαδήποτε συζήτηση υπάρχει για λύση δύο κρατών. μόνο η ομοσπονδία μπορεί να αποτελέσει διέξοδο ε, στη λύση αυτού του μεγάλου προβλήματος. σας καλώ σε αλληλεγγύη απέναντι στον κυπριακό λαό και καλώ και τους κύπριους σε αλληλεγγύη απέναντι σε όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν άλλοι λαοί στην ευρώπη. ευχαριστώ. Σας ε, επέτρεψα να μιλήσατε παραπάνω γιατί μας προσχεθήκατε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία σας ομιλία. Ο κύριος ε, Κάρβερ, για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, την προηγούμενη εβδομάδα ε, είδαμε σκάφη, σκάφη στην Μαύρη Θάλασσα να πλησιάσουν στο Νοβορσίσκ. Αυτή η περίπτωση ε, έδειξε επίσης ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ε, έχει τις ε, δικές του σκέψεις σχετικά με το αμυντικό σύστημα και τους S-400. Παρά λοιπόν τις απειλές και τις διαδικασίες που έχουν τρέξει στις ΗΠΑ, Πολιτείες. Βλέπουμε ότι εδώ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ρητορική Πολλοί αναφέρονται σε μια ενοποιημένη Ευρώπη, σε ενωμένε αμυντικέ δυνάμει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ το μόνο που ελπίζω είναι ότι μετά τι εκλογέ η πλειοψηφία να απορρίψει όλα αυτά τα μάντρα και να κατανοήσει ότι το ΝΑΤΟ είναι ο μόνο χώρο ειρήνη στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, κατά την άποψή μου ε, δεν θα πρέπει να έχουμε αυτή την προσπάθεια της στρατιωτικοποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και αυτό είναι εξίσου επικίνδυνο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάρβερ. Ο κύριος Μποργέτσιο, ένα λεπτό. Εμείς έχουμε στηρίξει τη θέση ότι είναι πολύ επικίνδυνο να υπάρχει ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η δική μας Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δεχτεί μια χώρα που δεν έχει τις προοπτικές να ενταχθεί σε αυτή. Όχι διότι θεωρούμε ότι η Τουρκία δεν ανήκει στην Ευρώπη. Όχι, δεν είναι έτσι. Σίγουρα ένα κομμάτι σημαντικό της Τουρκίας ανήκει στην Ευρώπη. Ε, βεβαίως, ε, μην ξεχνάτε ότι και κατά τη διάρκεια του φασισμού, ε, τότε το 1932 είχαν προσκαλέσει και την Τουρκία στη συνέλευση. Τότε όμως ήταν μια λαϊκή Τουρκία, δεν ήταν η σημερινή Τουρκία του Ερντογάν που έχει όνειρο το Ισλαμικό Χαλιφάτο. Η σημερινή Τουρκία ε, μας προκαλεί φόβο. Είναι εκείνη που αφήνει και τους τρομοκράτες να μπαινοβγαίνουν. Η Τουρκία είναι μια χώρα που χαρακτηρίζεται από ανομία και έχει διαλέξει ακριβώς αυτό τον δρόμο. Δέχεται όλους αυτούς τους ε, πρόσφυγες από τη Συρία και πολλούς τρομοκράτες. Γι' αυτό εγώ τη συγχαίρω για την υποκρισία της. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους 150 δημοσιογράφους που είναι έγκλειστοι στις φυλακές και αυτό πραγματικά είναι όνειδος. Ο κ. Επιτίδιος. Απεικονίζει την πραγματική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Δηλαδή, παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συλλήψεις και βασανιστήρια αντιφρονούντων και μη χειραγώγηση της δικαιοσύνης διώξεις αντιφρονούντων στο εξωτερικό και κατάργηση της ελευθερίας του τύπου. επίσης επισημαίνει την μη αναγνώριση της κυπριακής δημοκρατίας από την τουρκία το ότι δεν της επιτρέπει να εκμεταλλεύεται τους πόρους στην οικονομική της ζώνη και επίσης διότι παραβιάζει συνεχώς τον εναέριο χώρο της ελλάδος και τα χωρικά ύδατα και επιπλέον προκαλεί και δεν αναγνωρίζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου. όλα αυτά που ανέφερα δεν είναι απλές διμερείς διαμάχες μεταξύ της τουρκίας και των γειτόνων της είναι μια ευθεία παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου και προκειμένου να υποχρεωθεί η τουρκία να συνετιστεί θα πρέπει να διακοπούν άμεσα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσεις για την τελωνειακή ένωση και η χρηματοδότησή της. είναι απαράδεκτο να χρηματοδοτεί η ευρωπαϊκή ένωση την αγορά τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης ε, κόμπρα δύο από την τουρκία. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Δέχομαι την προοπτική που προέβαλε η κυρία Ζόμερ και ως προς την Κάτι Πύρη την είχα συμβουλέψει εδώ και δύο χρόνια αλλά το Συμβούλιο μας αγνόησε, αγνόησε τις υποδείξεις μας. Δεν θα πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία θέλγονται από τη στάση του Ερντογάν και μέσα στα πλαίσια της Προεδρίας. Η Τουρκία πολλές φορές αποτελεί δέλεαρ. Τι είδαμε τι έγινε στο Σαράγεβο. Ε, δηλαδή η Τουρκία ε, είναι ε, μία αρνητική δύναμη για ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά δελεάζει άλλα. Αυτή είναι η ιστορία μας. Όμως η Τουρκία θα πρέπει να αποσυρθεί από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Φλέκενστάιν για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων στην Τουρκία ε, δέχονται, είναι αναγκασμένοι να δεχτούν την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων. Έχει έρθει λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπέμψει ένα σαφές μήνυμα και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις που έτσι κι αλλιώ έχουν κολλήσει να πάψουν να συνεχίζονται. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι εγκλειστοί στις φυλακές και περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου χωρίς δίκαιη δίκη. Το αίτημα του Ευρωπαϊκού, Δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξει πλήρη πλήρης ε, αναστολή των ε, διαπραγματεύσεων είναι πολύ σημαντική γιατί τελικά είχαμε ζητήσει και παλαιότερα να ε, συνεχιστούν διαπραγματεύσεις μόνο αν υπάρξουν μεταρρυθμίσεις. Η επίσημη διακοπή πρέπει να λάβει χώρα έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής. Εμείς λέμε να ανασταλούν οι διαπραγματεύσεις, όχι να διακοπούν, όχι να πάψουν να υπάρχουν η πόρτα είναι μισόκλειστη. Παρά το αυστηρό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι σημαντικό στρατηγικό τέλο και δεν πρέπει να τη κλείσουμε κατά μουτρα την πόρτα. Βεβαίω, οι συζητήσει ε, με την τουρκική κυβέρνηση, στι συζητήσει αυτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε την κοινωνία των πολιτών. Τώρα ακριβώ ε, τι χρειάζεται, τώρα χρειάζεται την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα σταματήσει να ζητάει δικαιοσύνη για τον Ντεμιρτάς αλλά και για όλους τους άλλους έγκλειστους που βρίσκονται άδικα στις φύλακες. Βίστησεν παρακαλώ για ένα λεπτό. Η Τουρκία ιστορικά και πολιτιστικά είναι μια χώρα η οποία ανήκει στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό το ότι το κοινοβούλιο αυτό ε, κατάρτισε μία ε, έκθεση που ασκεί κριτική στην Τουρκία. Ε, δεν μπορούν να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις. Η Τουρκία εδώ και αρκετό καιρό καταδεικνύει ότι διολυσταίνει περισσότερο προς την κατεύθυνση του Ισλαμικού κράτους και με την ε, επιρροή της ε, Τουρκίας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε την ε, κατοχή της Κύπρου. Μην ξεχνάμε και πώς φέρεται η Τουρκία σε Τούρκους που ζουν σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Τώρα πρέπει να τους πούμε φτάνει πια. Να καταλάβουν δεν θα γίνουν ποτέ μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παύλα και τελεία. Ευχαριστώ κύριο Σαλή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κυρία Πύρη, αγαπητοί συνάδελφοι, το τελικό κείμενο τη έκταση του 2018 για την Τουρκία δεν μα βοηθά για να έχουμε ένα επικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και του στρατηγικού μα εταίρου. Η αναστολή τη ε, διαδικασία διαπραγμάτευση είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Πριν την τελική απόφαση που θα πάρουμε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τι πρόσφατε πρόοδου που δημιουργήθηκαν στην Τουρκία. Το Δεκέμβριο του 2018, η πέμπτη συνάντηση τη ε, ε, ομάδα δράση για τι μεταρρυθμίσει έλαβε χώρα στην Άγκυρα και είπαμε και υπόθηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει την προσπάθειά τη ε, έτσι ώστε να φτάσει στα ευρωπαϊκά πρότυπα παρά τα εμπόδια. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία εποπτείας ε, ε, του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ο υπουργό δικαιοσύνη θέλει να προχωρήσει σε μια στρατηγική μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη από κοινού με το Συμβουλίο της Ευρώπης και τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μπορέσουν να ενισχυθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην υπάρχουν παραβιάσεις τη σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η, μια αναστολή ή διακοπή τη διαπραγματική διαδικασία θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην Τουρκία. Αυτό φάνηκε στην συνεδρία τη ομάδα εργασία στην Άγκυρα. Υπό, υπό το φω των επόμενων ευρωεκλογών ε, στην, ε, θα πρέπει απέναντι στην Τουρκία να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι μηνύματα στέλνουμε προ του ε, εκλογεί. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Σολέ για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ο κύριο Σολέ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα ψηφίσουμε για την επίσημη αναστολή των διαπραγματευτικών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Το 2004 είχαμε ψηφίσει υπέρ του να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει. Από τότε έχουν γίνει πολλά χρόνια, από τα τελευταία 15 χρόνια. Οι σχέσει μα ήταν δύσκολε, συχνά, όμω ε, το αδιέξοδο αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει εάν είχαμε χρησιμοποιήσει το πλαίσιο προσχώρηση τη προσχώρηση, τη ένταξη και αν η Τουρκία βεβαίω είχε συνεχίσει το δρόμο προς περισσότερη δημοκρατία και προ τι μεταρρυθμίσει. Δυστυχώς η κατάσταση στην Τουρκία έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, βασικέ ελευθερίε. όλα αυτά βρίσκονται υπό σημαντική πίεση. Η πρόσφατη απόφαση που ζητάει δίκη η Σόβια του κυρίου Καβαλά είναι ένα από τα χιλιάδε παραδείγματα του τελευταίου διαστήματο. Βεβαίω η αναστολή της διαπραγματευτική διαδικασία στην Τουρκία δεν είναι λύση. Για να μπορέσει να μείνει ζωντανή η προοπτική τη δημοκρατία στην Τουρκία, ε, σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι λογικέ ελευθερίε, θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτέ τι πόρτε. Αν όχι για το παρόν, τουλάχιστον για το μέλλον. Αν όχι για εμά, τουλάχιστον για εκείνου στην Τουρκία, για του ανθρώπου, εκείνου που παλεύουν για ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη. Το να κλείνουμε την πόρτα και κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή. Η κυρία Μίχελς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Ερντογάν το αποτυχημένο πραξικόπημα το αποκάλεσε δώρο του Θεού. Οι ε, συνέπειε αναφέρονται στην έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Τουρκίας. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που έκανε το δώρο στην ε, Τουρκία. Επειδή υπάρχουν οι πρόσφυγες, για το λόγο αυτό συγκαλύφθηκε η δίωξη της αντιπολίτευση και υπήρξε και σιωπή στην περίπτωση της εισβολή στο Αφρίν. Εν τω μεταξύ η Γερμανίδα βουλευτή Ανασούκα απειλείται με τιμωρία τεσσάρων ε, ετών. Ε, αυτά είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η Τουρκία και κατά τα άλλα θέλω επίσης να επισημάνω ότι η δίωση η κατάσταση των γυναικών είναι εκείνη που υποφέρει πάρα πολύ από το καθεστώς Ερντογάν. Οι γυναίκες πρέπει να είναι αόρατες, να μην εκφράζουν την άποψή τους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε, ε, να αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε αν ε, δεχθούμε την αναστολή και ε, δεχθούμε σιωπηρά αυτή την στάση. Αυτό θα ήταν καλύτερο γιατί η Τουρκία δεν είναι μόνο Ερντογάν είναι η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών. Και αυτοί όλοι χρειάζονται τη δική μας τη φωνή. Θα δεχτείτε μία μπλε κάρτα από το συνάδελφό μας που κάθεται εκεί ψηλά από τον κύριο Σρόιντοβα. Κυρία Μίχελς, θα δεχτείτε την μπλε κάρτα από την κυρία Στρόιντοβα. Πολύ ωραία. Συνάδελφε, σ' άκουσα πολύ προσεκτικά κατ' ουσίαν μίλησες για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντάλλαξε την έλλειψη ελευθερίας στην Τουρκία με ε, άλλα δικά μας, με δικές μας απαιτήσεις αλλά δεν είναι αλήθεια. Εμείς δεν παραμένουμε σιωπηροί. Εμείς ε, έχουμε ψώσει τη φωνή μας ε, για τους έγκλειστους φυλακές. Η δική μας η αντιπροσωπεία μίλησε για τους πολιτικούς κρατούμενους. Ξέρετε τι ακριβώς λέτε. Συνάδελφε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε μια κατάσταση όπου όλες οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν ότι όσον αφορά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αυτή η συμφωνία μας κατέστησε εκβιάσιμους. Εγώ αυτό ακριβώς είπα, ότι μπορούμε πλέον να εκβιαστούμε. Ο Ερντογάν μας εκβιάζει εδώ και μήνες και χρόνια θα έλεγα, μας εκβιάζει κατά σύστολο τρόπο και νομίζω ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να σιωπούμε και αυτό το πρέπει να το επισημαίνουμε, όπως και όλα τα άλλα τα οποία έχουμε επισημάνει ή πρέπει να επισημάνουμε σε διάλογο που θα έχουμε με το καθεστώς του κ. Ερντογάν. Ο κ. Καστάλντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτή η συζήτηση γίνεται μια ιδιαίτερα σκόπιμη στιγμή. Έχουν απελαθεί τρεις Γερμανοί ρεπόρτερ από το τουρκικό έδαφος. Νομίζω ότι η Τουρκία διώκει τους δημοσιογράφους τόσο όσο καμία άλλη χώρα ανά τον κόσμο. Και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα ως προς τα ΜΜΕ. Η στάση του Σουλτάνου είναι αμήλικτη. Για να μην μιλήσουμε για άλλες κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Τουρκία συνεχίζει να είναι μια χώρα υποψήφια για προσχώρηση χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε καν να είναι δυνατόν. Η εισηγήτρια κάτι Πύρη διαχειρίστηκε με μεγάλη σύνεση αυτό το θέμα αλλά ήδη από το 2016 είχαμε ζητήσει να ανασταλούν οι διαπραγματεύσεις επίσημα. Αλλά μάταια ήταν αυτά τα λόγια, γιατί η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Συμβουλίου, το οποίο δυστυχώς καρκινοβατεί. Τα πράγματα δεν θα αλλάξουν από μόνα τους. Είμαστε υποκριτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το στρατηγικό γεωγραφικό ρόλο της Τουρκίας, αλλά δεν μπορούμε να μην στυλιτεύσουμε την στάση της. Η Τουρκία δεν έχει καμία αξιοπιστία. Θα πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Κάτι τέτοιο δεν βοηθά ούτε εμάς, ούτε τον τουρκικό πληθυσμό που κάποια στιγμή θα ζητήσει την δική μας λογοδοσία. Ο κύριος Κολομπιέ για ένα λεπτό. Η κυρία Πύρη δεν μπορεί να μην δεχτεί την πραγματικότητα. Η κατάσταση στην Τουρκία είναι άκρος ανησυχητική. Όμως η έκθεση Πύρη προβαίνει σε μια αρνητική ανάλυση της κατάστασης χωρίς όμως να μιλά για την προοπτική προσχώρηση. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολιτισμικούς λόγους. Παρόλο που εκτιμούμε τον τουρκικό λαό. Θεωρούμε ότι η Τελωνιακή Ένωση θα αντιστρεφόταν στα δικά μας συμφέροντα τι θέλουμε, περισσότερες φυλακίσεις, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι θέλουμε πλέον. Θα ήθελα, συνάδελφοι, να υπερψηφίσετε το εναλλακτικό ψήφισμα του ΙΕΝΕΦ που ζητά τη μόνιμη αναστολή των διαπραγματεύσεων, την ακύρωση δηλαδή.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 η αστική τάξη της τουρκίας εντείνει την επιθετικότητά της γκριζάροντας χωρικά ύδατα και ένα αέριο χώρο με διαρκείς παραβιάσεις παράνομες ναύτες στρατιωτικές ασκήσεις και απειλές ενώ η κυβέρνηση σύριζα εμπλέκεται στους ανταγωνισμούς ως σημεοφόρος των ευρωατλαντικών σχεδιασμών στην αντιπαράθεση με τη ρωσία προσπαθεί να ξεπλύνει τον επικίνδυνο ρόλο των ηπα νατο ευρωπαϊκής ένωσης και καλλιεργεί τον εφησυχασμό. Όσε επικριτικέ διατυπώσεις για τον ερντογάν και αν περιλαμβάνουν οι εκθέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζονται από το δεδομένο ρόλο στρατηγικού εταίρου που αποδίδουν στην τουρκία φωτογραφίζοντα την ευρωνατοϊκή διευθέτηση σε αιγαίο για συνεκμετάλλευση καθώ και το διχοτομικό σχέδιο στην κύπρο προκειμένου να μοιραστεί η πίτα τη ενέργεια. προκαλούν δε μεγάλα ερωτηματικά θολές αναφορέ στην έκθεση για επίλυση διμερών διαφορών που εκκρεμούν για μη διευθετημένες νομικέ υποχρεώσει και ανεπίλητε διαμάχες με στους άμεσους γείτονες όσον αφορά χερσαία θαλάσσια σύνορα και ένα αέριο χώρο. η λαή επιβάλλεται να είναι σε τιμότητα με πάλι ενάντια στον εθνικισμό και τα υπερελιστικά σχέδια ευρωπαϊκής ένωσης νάτο και αστικών τάξεων. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κάζα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. με τη σημερινή της ε, ε, κυβέρνηση απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από την ενταξιακή προοπτική η Τουρκία. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική δημοκρατία αν δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Ε, βλέπουμε την κατάσταση στην Τουρκία με την περίπτωση των δημοσιογράφων. Βλέπουμε τι γίνεται με την ερευνητική δημοσιογραφία και τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο που είχε κάνει μία αναφορά για Paradise Papers και τώρα ε, κινδυνεύει να καταδικαστεί ε, σε πολλαπλά πρόσθεμα και σε 13 ε, μήνες κάθυρξη. Είναι μία ε, νέα μητέρα και αν ε, η ποινή της εκτελεστή θα χωριστεί από το μωρό της. Πρόκειται για μια ομή βάναυση άκαρδη κυβέρνηση. Αξίζει καλύτερα η Τουρκία. Γι' αυτό καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σας ζητώ να αναλάβετε δράση άμεσα, να απαιτήσετε να ε, πέρσουν οι κατηγορίες κατά της Πίλεν Ούλκε, αυτής της δημοσιογράφου. Κύριος Κύρκος δίθεν αναστολή αλλά ουσιαστικά οριστική διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την τουρκία. το θέλει μεταξύ άλλων εμφατικά ο κύριος βέμπερ που θεωρεί ότι η τουρκία δεν έχει θέση στην ευρωπαϊκή ένωση ό,τι και να κάνει έστω και είκοσι χρόνια αργότερα. η συμφωνία siemens και deutsche bahn των τριάντα δύο δισεκατομμυρίων για τους τούρκικους σιδηρόδρομους μας δείχνει το προνομιακό πεδίο σχέσεων ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας που κάποιοι οραματίζονται χωρίς φυσικά τα ενοχλητικά κριτήρια της κοπενχάγης το θέλουν όμως κι άλλοι ως τιμωρία του προέδρου ερντογάν για την απαράδεκτη παραβίαση του κράτους δικαίου. όμως όλοι οι δημοκράτες στην τουρκία μέσα και έξω από τις φυλακές και ο καβαλά και ο ντεμιρτάς όλα τα πολιτικά κόμματα σε μια σπάνια στιγμή σύμπνοιας ζητούν να μην σκοτώσουμε το ευρωπαϊκό όνειρο της χώρας τους. εμείς ξέρουμε καλύτερα ε! business as usual και δίθεν ηθικό πλεονέκτημα χέρι με χέρι ακυρώνουν την ευρωπαϊκή προοπτική ενό λαού τη γειτονιά μα αλλά και το μόνο εργαλείο θεσμική μα παρέμβαση εκεί όπω σωστά υποστηρίζει και η ελληνική κυβέρνηση. ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε κύριο Φανόρντεν για ένα λεπτό. Ναι, πάντοτε θεωρούσα ότι θα πρέπει να έχουμε κοντά μας την Τουρκία. Να την έχουμε από κοντά πιο σωστά γιατί τώρα βλέπουμε ότι ό,τι προσπάθεια προσχώρηση ή ένταξη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε γίνει ω τώρα ήταν ευνοϊκή και για την Τουρκία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερα να κανεί να ταξιδεύει, λέει κανείς, παρά να φτάνει στον προορισμό του. Αυτό το ταξίδι έχει κρατήσει 15 χρόνια. Κάποιοι θα λέγανε και 30 ίσω. Ε, και τώρα ε, προσθέτουμε ε, στην ε, ήδη δυσάρεστη κατάσταση κάτι ακόμα χειρότερο. Γιατί να αναστείλουμε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να δημιουργήσουμε εχθρική διάθεση στου γειτονέ μα. Κύριε Μπαρνιέ, σημειώστε τα. Μέσα στα χρόνια βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει κάνει κάποια πρόοδο, ε, σε κάποια θέματα πάλι όχι. Ένα θέμα ήταν πάντοτε η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για τις δημοκρατικές αξίες, αγνοεί όμως την κατάσταση στο 1 τρίτο του νησιού, που εφόσον θέλουμε να διατίθεται στο λαό του, της νήσου θα πρέπει να εκπροσωπείται και εδώ και θα έπρεπε να έχουν και ε, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης καθεστώς παρατηρητών οι τουρκοκυπροί. Ο κύριος Μό, ήταν λεπτό. Για μια ακόμη φορά μιλάμε για την ε, ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην, την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι για το οποίο θα έπρεπε να μιλάμε είναι Ισλαμικό κράτος έχει το χαλίφ του Βοσπόρου στο πιδάλιο της χώρας και δεν έχει τίποτα κοινό με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν ανήκει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δική μου ομάδα πολλές φορές έχει ζητήσει όχι απλά το προσωρινό πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αλλά την οριστική τους κατάσταση κατάργηση, ακύρωση, χωρί καμία άλλη προθεσμία. Έχουμε μια νέα ε, ευκαιρία γιατί είπε και ο Βέμπερ την εβδομάδα ότι αυτό ε, εάν γίνει πρόεδρο τη Κομισιόν ε, θα τερματίσει τι προταξιακέ συνομιλίε. Γιατί περιμένετε, γιατί περιμένετε τσεντεου τσέσου αγαπητέ Βέμπερ, γιατί το κάνετε από τώρα αυτό. Έχουμε την τροπολογία 17. Ζητάμε με αυτήν οριστική πάυση των πρωταξιακών διαπραγματεύσεων. Δεχτείτε τι. Και ακόμη και πριν τις ευρωεκλογές Καλό είναι να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πραγματικά ε, θέλουμε να διακόψουμε οριστικά αυτέ τι ενταξικέ διαπραγματεύσει. Μάρουση για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μπροστά μας ένα κείμενο, πολύ καλογραμμένο, ε, αλλά δεν είναι λογοτεχνικό κείμενο. Δεν ε, ταιριάζει η γλώσσα αυτή στην σκληρή πολιτική πραγματικότητα η ε, πολιτική είναι η τέχνη του να μπορεί κανείς ε, να δημιουργήσει κάτι, να ασκήσει την δύναμή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσεται πάρα πολύ βραδέως, ε, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με την Τουρκία, η οποία όλο και αναπτύσσεται και όλο και πιο ανελέητα στρέφεται κατά όλων της των αντιπάλων το να εκφράζουμε την χαρά μας για τις σχέσεις της Τουρκίας με τον ΝΑΤΟ είναι πραγματικά δείγμα μεγάλης αφέλειας. Οι ασκήσεις ε, των ε, τουρκικών και ρωσικών δυνάμεων, η αντιοαεροπορική ε, πύραυλη, ε, τα νέα αυτά πυραυλικά συστήματα που αποστέλλονται στην Τουρκία. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάνει μια προσπάθεια να νοικοδομήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συναδεινός για ένα λεπτό. Πριν δύο χρόνια από αυτό το βήμα είχα επισημάνει τον ύπουλο τρόπο με τον οποίο η Τουρκία του Ερντογάν κλείνει συμφωνίε. Είχα καταδικάσει την προσπάθεια εξαγορά τη Τουρκία με επακτολό δισεκατομμυρίων ευρώ για λύση του μεταναστευτικού. Εκδιώχθηκα κατά παράβαση του κανονισμού από την αίθουσα από τον τότε πρόεδρο σουλτ. δύο χρόνια μετά η ένωση σπατάλησε κοντά πέντε δι όμως η ευρώπη πλημμύρισε σε λαθρομετανάστες. ο σουλτ πήγε σπίτι του αποτυχάνοντα τη γερμανική πολιτική σκηνή όμω το καταστροφικό του πέρασμα παραμένει. ο βέμπερ υιοθέτησε τη ρητορική μου και αυτό δεν με κάνει απλώ ικανοποιημένο αλλά κυρίω δικαιωμένο. βέβαια δεν βλέπω του ευρωβουλευτέ τη Ελλάδο που ανήκουν στο ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα να κατηγορούν τον βέμπερ για ρατσισμό όπω έκαναν στη δική μου περίπτωση νομοτελειακά στι επερχόμενε εκλογέ η ευρώπη θα γυρίσει σελίδα. οι πατριωτικέ ευρωσκεπτικιστικέ δυνάμει θα σαρώσουν τι απάτριδε διεθνιστικέ και εθνομηδενιστικέ τάσει. ευχαριστώ. Eh, με συγχωρείτε, Δεν πειράζει. Θα ξεκινήσω τώρα με το ένα λεπτό μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, την εισηγήτρια μάλλον, συγγνώμη, για την έκθεσή της, την κυρία Πύρη. Δεν είναι καθόλου απλό να πετύχει κανείς μια ευρεία πλειοψηφία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σε αυτό το σώμα και όμως το πετύχατε εσείς και γι' αυτό συγχαρητήρια. Ε, είναι εντονότερη στην έκφρασή της αυτή η έκθεση από ό,τι συνηθίζεται με τέτοιες εκθέσεις που απλώς ε, καθησυχάζουν και καταπραίνουν τα πνεύματα. Εδώ λοιπόν ε, αυτό που λέει η έκθεση είναι ότι θα πρέπει οι διαπραγματεύσει να σταματήσουν. Ε, και αν ακούσετε τι λένε και οι συνάδελφοι, ε, θα ακούσετε ότι ε, χρόνο το χρόνο η Τουρκία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική εταιρική σχέση για να αντικαταστήσουμε αυτή την πορεία. Θα πρέπει να βρεθεί κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε στην κατάρκηση των διαπραγματεύσεων. Και θα έλεγα ότι κρίμα που η ίδια σα η τροπολογία, η τροπολογία 21, λέει να αναστείλουμε τι διαπραγματεύσει. Αλλά μην ανασυχείτε γιατί η ευρωπαϊκή σα υποψηφιότητα παραμένει ενεργή. Είναι περίεργο. Ευχαριστούμε. Και πάλι συγγνώμη. Απλώς κάτι κοίταζα στα έγγραφα και ξέρω πολύ καλά το όνομά σας, αλλά έγινε ένα μπέρδεμα προσωρινά. Η κυρία Λόπες, για ένα λεπτό. Ο κύριος Λόπες, συγγνώμη. Για ένα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγητρία, την Κάτι Πύρη για τη δουλειά της, ε, όχι μόνο τη φετινή, πέντε χρόνια ε, ακούραστα, άοκνα εργάστηκε για την Τουρκία και δεν ήταν πάντα εύκολο το έργο της σήμερα ε, για νιωστή φορά ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προειδοποιούμε τον Ερντογάν για τη θεσμική υποβάθμιση των τελευταίων ετών, μια επιδείνωση ιδίω μετά το πραξικόπημα πάρα πολύ έντονη. Βλέπουμε ότι αποδεκατίστηκε η δημόσια διοίκηση, ότι παραβιάζονται συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν γίνονται σεβαστέ οι μειονότητε. έχουμε κρατήσει ε, των δημοσιογράφων καθημερινά και αυτό το οποίο έγινε η σταγόνα που έκανε να ξεκυλήσει τελικά το ποτήρι ήταν οι συνταγματικέ μεταρρυθμίσει που ουσιαστικά έχουν μεταμορφώσει την ταυτότητα τη Τουρκία. Αντί να είναι σύγχρονη, μοντέρνα χώρα, είναι μια μονολυθική χώρα. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα όμω. Ο Ερντογάν δεν είναι Τουρκία. Χρειάζονται λοιπόν διάβλη επικοινωνία. Ποιε και με ποιου όρου και προποθέσει. Πρώτον, εξυγχρονισμό ε, τη ε, Συμφωνία για την Τελωνιακή Ένωση και απελευθέρωση θεωρήσεων, ώστε να ξαναμπεί στο δρόμο του δικαίου η Τουρκία. Σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Θεοχάρου για ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο παρακαλούμε. My micro, please. It turn on now. Thank you. Is it okay? Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η έκθεση παραγνωρίζει πλήρως τις βασικές αρχές δικαίου για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και όχι μόνο υποστηρίζει αναλυθή γεγονότα αλλά ψεύδεται κατάφορα όταν αναφέρεται σε δίθεν συμφωνία που επετεύχθη στο κραν μοντανά. η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που εισηγείται η έκθεση ως λύση του κυπριακού δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης και οδηγεί σε εκτουρκισμό της κύπρου το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έχει ήδη βαρύτατη ευθύνη που αποδέχεται τα δεδομένα της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής του νησιού. η έκθεση απαλλάσσει την τουρκία κάθε ευθύνη για τη μη επίλυση του κυπριακού και δεν κάνει αποδεκτή την διασύνδεση αναγνώρισης της κυπριακής δημοκρατίας με την πρόοδο των ενταξιακών. για παράδειγμα πώς θέλετε επικαιροποίηση της, ε, της συμφωνίας τελωνειακής ένεσης όταν δεν έχει εφαρμοστεί η υφιστάμενη; η τουρκία απειλεί συνεχώ και εμπράκτο την κύπρο. η έκθεση αντιμετωπίζει τι απειλέ με ευχολόγια. θα καταψηφίσω την έκθεση επειδή περιέχει ψεύδι. ζητά να συνεχιστεί μια επικίνδυνη διαδικασία πλήρου κατάκτηση τη χώρα μου από την τουρκία νομιμοποιεί την κατοχή στηρίζει την ένταξη ενό δικτατορικού καθεστώτο στην ευρωπαϊκή ένωση. και βεβαίω για όσου θέλουν συνέχιση των ενταξιακών Συγγνώμη, ε, ένα λεπτό το χρόνο για το συντομότερο, για, σημαντικότερο για τη χώρα μου θέμα την κατοχή χώρα μου. Ναι, το καταλαβαίνω, λέει ο πρόεδρο. Όλοι έχουμε θέματα που μα είναι σημαντικά, αλλά λυπούμε ότι οι κανόνε είναι κανόνε πρέπει να του σεβαστώ. Αυτή είναι η δική μου υποχρέωση. Αλλά νομίζω παρόλα αυτά το μήνυμά σα ήταν απολύτω σαφέ. Ευχαριστώ, σαφές. Ευχαριστώ για την κατανόησή σα. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Αρνοτού για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώριζε επισήμω το καθεστώ υποψηφίου χώρα στην Τουρκία υποψήφια για την ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 20 χρόνια μετά έκθεση αυτή καλεί στην αναστολή των διαπραγματεύσεων. Και πάλι το Κοινοβούλιο όμω δεν λαμβάνει απόφαση. Ενώ θέλει να αυτοκολακεύεται με μια, ότι χρησιμοποιεί εκφράσει χωρί ε, χωρίς υποκρισία. Πότε θα περιμένουμε άλλα 20 χρόνια για να φτάσει η Τουρκία να πάρει απόφαση ότι θα είναι ποτέ μέλο. Ε, αντίθετα με του φιλευρωπαϊστέ, η γραμμή μα θα είναι πάντοτε σταθερή. Το 1986 ο Λαϊπέν έλεγε ήδη σε ένα λόγο ότι η Τουρκία δεν έχει καμία ευρωπαϊκή θέση, ούτε από τη γεωγραφική τη θέση, ούτε την ιστορία τη, ούτε τον πολιτισμό τη. Ακόμη και αν αυτό δεν αρέσει στου προαπιστέ μια πολυπολιτισμική Ευρώπη και αυτού που προασπίζονται όπω ο Εντρογάν και ο Σιράκ στην εποχή του, ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι ένα κλαμπ χριστιανών. Η Τουρκία έχει εξισλαμιστεί από την πτώση τη Κωνσταντινούπολη και ε, οι χριστιανοί ήταν πριν από 100 χρόνια ένα τέταρτο του πληθυσμού τη Τουρκία, σήμερα είναι μόνο 1%. Αυτή η τραγωδία και μόνο δικαιολογεί το να ζητήσουμε την οριστική διακοπή των διαπραγματεύσεων και όχι απλώ μια αναστολή. Ευχαριστούμε ένα λεπτό, κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Η Τουρκία είναι ο στρατηγικός μας εταίρος σε θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης. Φυσικά και πρέπει να καταγγείλουμε απερίφραστα την ε, ε, δίωξη των πολιτικών αντιπάλων ε, με το πρόσχημα της αντιτρομοκρατικής δράσης. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Το έχουμε ξαναζητήσει αυτό και πιστεύω ότι έχουν πραγματικά συμφέρον ε, οι Τούρκοι να ε, προωθήσουν μέτρα, ε, θέλουμε να συμμετέχουν ε, στο Εράσμος και σε άλλα προγράμματα. Δεν σημαίνει ότι είμαι υπέρμαχος της προσχώρησης της χώρας ε, στην Ένωση, αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική πρόοδο, την κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει την αναστολή των δεξιακών διαπραγματεύσεων να τη χρησιμοποιήσει ως ένα μοχλό για τη δημιουργία μιας νέας σχέσης που θα οδηγήσει σε διάλογο. Ευχαριστώ κύριο Παπαδάκης Δημήτρη Κύριε για Πρόεδρε, λυπούμε να παρατηρήσω ότι εξελίσσεται ένα θέατρο παραλόγου και μια προσπάθεια εξυπηρέτησης συμφερόντων. Κάποιοι μιλούν για διακοπή, αλλά την ίδια στιγμή προωθούν την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης. Δηλαδή, καμία υποχρέωση από πλευράς Τουρκίας, αλλά να εξυπηρετήσουμε τα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα και στις δύο πλευρές και σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και στην ίδια την τουρκία. αυτό θέλουμε; επιτέλους ας γίνουν ξεκάθαρα τα πράγματα. θέλουμε να έχει ευρωπαϊκό δρόμο και προοπτική η τουρκία μόνο αν σέβεται τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης. ας προβληματιστούμε τι έγινε μέχρι σήμερα με την πολιτική που ακολουθήθηκε; φυλαγίζει τούρκους πολίτες εξωστραγίζει ευρωπαίους δημοσιογράφους συνεχίζει να κατέχει το 40% της κύπρου και απειλεί καθημερινά την αποκλειστική οικονομική ζώνη ενός κράτους μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης. Ευχαριστούμε κύριο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, με τη σημερινή μου ομιλία συμπληρώνω 2.500 ομιλίες και παρεμβάσεις στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην παρούσα θητεία και θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι η ομιλία μου αυτή αφορά την τουρκία την τουρκία η οποία συνεχίζει παράνομα να κατέχει το 37% του εδάφους της κυπριακής δημοκρατίας την τουρκία που συνεχίζει τις απειλές κατά της ελλάδος και παραβιάζει τα ελληνικά χωρικά ύδατα και τον ελληνικό εναέριο χώρο την τουρκία η οποία αρνείται να συμμορφωθεί προς το διεθνές δίκαιο και να επιτρέψει στους έλληνες της δωδεκανήσου να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες τους και όλα αυτά παρότι η κομισιόν μετά από παρέμβασή μου έχει αναγνωρίσει ότι υφίσταται το θέμα για τις επωνομαζόμενες δωδεκανησιακές περιουσίες. μόνη λύση για να αναγκαστεί να συμμορφωθεί η άγκυρα είναι η επιβολή κυρώσεων διπλωματικών και οικονομικών κατά της τουρκίας. εδώ και τώρα άμεσος τερματισμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας και πάυση κάθε χρηματοδότηση από πλευράς ένωσης προς την τουρκία. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσόκα για ένα λεπτό. Η Λίγκα είχε πει όχι στην προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρώπη και θα συνεχίζει να το λέει. Γιατί. Γιατί είναι ένα εγχείρημα τρελό, εγκληματικό. Τι μπορούμε να Τι σκέφτεται κανεί, ότι μια χώρα που είναι 100% μουσουλμανική θα μπει στην Ευρώπη, θα καταστρέψει τελείω τη Δύση κάτι τέτοιο. Η Λίγα λέει όχι. Διότι ένα στου πέντε πολίτε, ένα στου πέντε Τούρκου, λέει ότι του αρέσει το Άιζη. 30 εκατομμύρια πρόσφυγες είναι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι έχουν παραβιαστεί με εγκληματικό τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα εις βάρος γυναικών, εις βάρος ανηλίκων. Για αυτούς τους λόγους θα συνεχίζουμε να λέμε διαρκώς και ε, με πείσμα όχι στην είσοδο τη Τουρκία στην Ευρώπη. Θα ήταν εγκληματικό να θέλουμε να συνεχίσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα που ήδη κόστησε 11 δι στου Ευρωπαίου πολίτε. Τα πετάξαμε από το παράθυρο για να, για να πιστούμε ότι μπορεί η Τουρκία να μπει στην ε, Ευρώπη. Η... Αυτά θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν σε πολίτε τη Ευρώπη και τη Ιταλία. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Αντέμοφ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, είναι σαφές για όλους μας ότι η πλήρη συμμετοχή της ε, Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι του παρόντος. Γι' αυτό το λόγο οι διαπραγματεύσει το 2005 είχαν ξεκινήσει χωρίς καμία εγγύηση ότι θα υπάρξει αισιοπέρας. Η Τουρκία αντιμετώπιζε, ήδη πολλά προβλήματα σε πολλούς τομείς, την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις αξίες. Όλα αυτά είναι μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και όμως τώρα θεσμικοί φορεί τη χώρα σε μεγάλο βαθμό και ένα μέρο του πληθυσμού δεν εγκρίνουν τόσα συμβαίνουν εκεί. Θα έπρεπε η ευρωπαϊκή πολιτική να ενθαρρύνει μεταρρυθμίσει για να προωθήσει τη δημοκρατία στην Τουρκία. Είναι σημαντική η Τουρκία και για την εξωτερική μας πολιτική, για την ασφάλεια, και την κοινή καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, είναι η σύσταση για την αναστολή των δημοκρατήσεων με την Τουρκία σωστή. Μήπως θα έπρεπε να μην γίνει μεγαλύτερο το χάσμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, αλλά ασφαλέστερο το σύνορό μας. Θα πρέπει να σκεφτούμε και τους Τούρκους πολίτες που είναι φιλευρωπαϊστές και ε, να μην οδηγήσουμε σε προσδοξισλαμισμό εξισλαμισμό και ριζοσπαστικοποίηση την χώρα. Φρόιντ, για ένα λεπτό. Είχα συγχαρεί προσωπικά την κυρία Κατυπήρη και δεν θα το επαναλάβω. Έχω χρηματίσει δημοσιογράφος για πολλά χρόνια και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της ε, ελευθεροτυπίας και δεν βλέπω στον ορίζοντα βελτίωση της κατάστασης. Έχουμε στη φυλακή δημοσιογράφου στην Τουρκία επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Είναι απαράδεκτο αυτό όπως και το ότι εκπρόσωποι ε, ξένου τύπου ε, χάνουν τα διαπιστευτήριά τους όπως το Τσεντεφ ή το Τάγκε Σπίγκελ, οι εκπρόσωποι αυτών των μέσων ε, και ε, επίσης ε, ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάθισε για μήνες ολόκληρες στη φυλακή χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ε, δεν θέλουν ε, την κυβέρνηση Ερντογάν. Όμω δεν θέλουμε να στραφούμε με την ε, αναστολή των διαπραγματεύσεων σε βάρο των πολιτών τη Τουρκία, αλλά σε βάρο τη κυβέρνηση Ερντογάν. Να καταστεί σαφέ ότι στηρίζουμε τι φιλευρωπαϊκέ και τι προοδευτικέ δυνάμει στην Τουρκία, ότι δεν του εγκαταλείπουμε. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριο Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε Τέλιτσκα. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Πύρη για την έκθεσή της. Βλέπω επιτέλους μια έκθεση για την Τουρκία που να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Δεν είναι ευρωπαϊκό κράτος η Τουρκία παρεμβαίνει για τον γειτονικών χωρών, όπως της Βουλγαρίας για παράδειγμα. Πρόκειται για παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα μιας άλλης χώρας η οποία είναι εντελώ απαράδεκτη και σε ό,τι αφορά τους ε, μουσουλμάνους στη Βουλγαρία και σε ό,τι αφορά την ε, απόπειρα ε, συγκρότηση πολιτικού κόμματος και επηρεασμού του πολιτικού βίου της Βουλγαρίας. Απαράδεκτα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα επιτρέψουμε. Γι' αυτό και επιμένω ότι θα πρέπει να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις και ελπίζω αύριο η ψηφοφορία αυτό το αποτέλεσμα να έχει. Έτσι ε, θα χρειαστεί ε, και από την πλευρά της Κομισιόν να δούμε να παίρνει την απόφαση να σταματήσει οριστικά. Κύριος Μακάλιστερ έχει το λόγο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, εξωτήμες κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι ακρογωνίω λίθος της δημοκρατίας, είναι προϋπόθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό ε, το εδάφιο 8 ε, της έκθεσης κάτι πύρη, διότι πραγματικά ε, δεν πρέπει να υπάρχουν δυσανάλογα μέτρα καταπολέμηση και περιορισμού της Ε, ε, και πρέπει να σας πω ότι Χρειάστηκε πολλοί ε, Γερμανοί ε, δημοσιογράφοι να αποχωρήσουν από την Τουρκία γιατί τους ε, πήραν την άδεια, τις διαπιστεύσεις τους, ανταποκριτές που εκφράζουν κριτική άποψη αντιμετωπίζονται ως τρομοκράτες, ως εχθροί της Τουρκίας. Αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Πραγματικά είναι κατάφερες παραβιάσεις κατά της ελευθεροτυπίας. Πόσο, ποτέ δεν θα σταματήσουμε και δεν θα αφιστούμε να τις καταγγέλουμε. Ο κύριος Μάμικη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τη συνάδελφα Κάτι Πύρη, την εισηγήτρια ε, μιας πολύ σημαντική έκθεσης. Επίσης θέλω να πω ότι με την αποχώρηση Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία γίνεται όλο και πιο σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας για την επίλυση του ε, προβλήματος ασφαλείας. Είναι ένας ε, παίκτη πολύ σημαντικός ε, για να βοηθήσει ε, να τερματιστεί η οκτάχρονη ε, σύγκρουση ε, στη Συρία και έχει στηριχθεί η διαδικασία της Αστάνα ρόλος του Ιράν, της Ρωσίας, της Τουρκίας είναι σημαντικός η Ρωσία και η Τουρκία απέτρεψαν την ανθρωπιστική καταστροφή με την εκεχηρία ε, για την οποία εργάστηκαν. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε ε, τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Είναι πολύ σημαντική η διαδικασία της Αστάνα για μια πιο ασφαλή Ευρώπη και για την αποτροπή επιθέσεων από ξένους μαχητές. Ευχαριστούμε ο κύριο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Διάβασα πολύ προσεκτικά την έκθεση, η οποία επικρίνει σοβαρά την Τουρκία. Και έχει και πάρα πολλέ ε, λεπτομερεί πληροφορίε για το τι πηγαίνει στραβά σε αυτή τη χώρα, για την απόπειρα του πραξικοπήματο το 2016 και το καθεξή. Εκεί όμω που δεν βλέπω να υπάρχουν αρκετά είναι τα συμπεράσματα. Ε, δηλαδή, να σταματήσουμε τη χρηματοδότηση ε, τη Άγκυρα για το διευκόλυνση των προσφύγων, το δεύτερο μέρο. Ήδη έχει μειωθεί ένα μερίδιο μόνο του συνόλου που η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει στην Τουρκία, αλλά η βοήθειά μας δεν έχει βοηθήσει. Ε, η βοήθειά μας μάλλον δεν έχει δώσει αποτέλεσμα, γιατί ε, η Τουρκία ούτω ή άλλω υποστηρίζεται τι ΗΠΑ. Δεν χρειάζεται λοιπόν απλώ να αναστείλουμε τι διαπραγματεύσει. πρέπει να τι διακόψουμε πλήρω. Η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει ποτέ μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Τελωνιακή Ένωση θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα. Ε, γι' αυτό λοιπόν νομίζω το μήνυμα του Συμβουλίου είναι το μήνυμα του Συμβουλίου είναι λανθασμένο. Δεν μπορεί να έχουμε μια τελωνιακή ένωση και να επιτραπούν όλα τα υπόλοιπα. Θα πρέπει ε, αυτό να αναφέρεται ξεκάθαρα στην έκθεση. Ευχαριστούμε, Χριστοφόρο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι στα θέματα τη Τουρκία κρίνεται η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουμε να προασπιστούμε τι ευρωπαϊκέ αρχέ και αξίε. Και αυτέ θα μπορέσουν να προασπιστούν εάν η Τουρκία υποχρεωθεί επιτέλου να σεβαστεί και τα ψηφίσματα και τι εκθέσει. από τη στιγμή που δεν σέβεται τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε εμεί οφείλουμε να αντιδράσουμε και η μοναδική αντίδραση όταν η τουρκία παραβιάζει αρχέ και αξίε στην κατεχόμενη κύπρο από τα τουρκικά στρατεύματα όταν παραβιάζει την κυπριακή ναό όταν προκαλεί την ελλάδα και την κύπρο χώρε μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση μία είναι η αντίδραση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου εάν δεν υλοποιήσει αυτά που καταγράφονται στην έκθεση να υποχρεωθούμε να παγώσουμε την προενταξιακή βοήθεια τη τουρκία. δεν ρωτήσαμε κανέναν ευρωπαίο πολίτη εάν θέλει να δίνει έστω και έναν ευρώ στην τουρκία σήμερα και οφείλουμε να το πράξουμε γιατί μόνο και μόνο έτσι η τουρκία θα συμμορφωθεί επιτέλου σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε και ποτέ δεν συμμορφώθηκε είναι αδιανόητο να υπάρξει αναβάθμιση τη τελωνειακή ένωση χωρί αναγνώριση τη κυπριακή δημοκρατία χωρί να σπάσει το αδιέξοδο των κυπριακών που παρά τη καλή θέληση του προέδρου τη κυπριακή δημοκρατία η τουρκία και ο ερντογάν παραμένουν αδιάλακτοι και προκλητικοί. ευχαριστώ πρόεδρε Επίτροπε δεν ξεχνάει το σημαντικό ρόλο που έχει η Τουρκία στην απόκρισή μα στην ε, μεταναστευτική κρίση και το τι συμβαίνει στον πόλεμο στη Συρία. Εν τω μεταξύ όμω αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να παραμένει μάλλον ε, να εμένει σε μια υποκριτική στάση που εμποδίζει να προχωρήσουμε. Ξέρουμε την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία, τι φυλακίσει που είναι εκατοντάδε, τις θεωρήσει που δεν δίνονται, τι πλατφόρμες τα ψηφιακά μέσα που ε, δεν επιτρέπονται, το ίδιο και στα κοινωνικά δίκτυα. Θα πρέπει από την άλλη όμω να θυμόμαστε ότι τα ίδια αυτά άτομα υπολογίζουν τη δική μα βοήθεια. Η κατάσταση είναι κακή και ήταν και από καιρό κακή. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει μια γέφυρα συνεννόηση με την Τουρκία μέσω διπλωματικών οδών. Θα πρέπει ο στόχο τη προσχώρηση τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση